Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ostern allerseits. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλό Πάσχα. Αρχίζει η συνεδρίαση τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Έκτακτη συνεδρίαση, λυπάμαι, ήταν όμω αναγκαίο για να συζητήσουμε διάφορα θέματα και γι' αυτό λοιπόν ήταν πάρα πολύ σημαντικό να συνεδριάσουμε από κοινού. Προβλέπεται επίσης και συνεδρίαση των συντονιστών και περνάμε στην ημερήσια διάταξη. Είναι πολύ σύντομη αλλά πολύ σημαντική. Ε, δεν υπάρχουν επιθυμίες για να αλλάξει η ημερήσια διάταξη. Εγκρίνεται λοιπόν. Τώρα σε ό,τι αφορά το γλωσσικό καθεστώς ε, το έχετε μπροστά σας και επίσης μεταδίδεται ζωντανά από το διαδίκτυο. Περνάμε στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης για τους δημοσιονομικού κανόνες. Έχω κάποια καλά νέα. Στις 27 Μαρτίου καταφέραμε να έχουμε μία συμφωνία για τα επίμαχα άρθρα, ε, το 182 για παράδειγμα, και αποφασίσαμε, ε, συμφωνήσαμε μάλλον, ε, να υπάρχει προθεσμία τριών μερών για τη δημοσίευση. Μετά τα άρθρα 6 58, 62, 67, 72, 200 και 256 έως 260 θα τεθούν σε σχέση από 1η Πρώτου του 2019. Μετά σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους θα, η ισχύ θα είναι τρεις μέρες μετά τη δημοσίευση. Τώρα, γιατί θέλουμε να εστιάσουμε ιδιαίτερα σε αυτά τα σημεία, γιατί κάθε θεσμικό όργανο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει ε, τους ε, δημοσιονομικούς κανόνες σύμφωνα με τις δικές του ανάγκες και αυτό θα είναι πιο εύκολο μάλιστα ενώπιον των ε, ευρωεκλογών, διότι διαφορετικά θα ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Πιστεύω πως έχουμε λοιπόν καταλήξει σε μια λογική και σωστή λύση και αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τον ε, τριμερή διάλογο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εδώ άλλη μια φορά όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτόν για την καλή συνεργασία. Τώρα σε ό,τι αφορά το κείμενο και το οποίο θα περάσει στην Κοροπέρ θα ψηφιστεί στην Επιτροπή μας σύντομα. Θα ήθελα εδώ να συγχαρώ τον συνεισηγητή κύριο Ashworth να σας αναφέρω τα κυριότερα σημεία. Δεν υπάρχει αναφορά σε καταπιστεύματα, δεν υπάρχουν καταπιστεύματα λοιπόν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διατηρείται η αρχή του non-profit, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Υπάρχουν, δεν Υπάρχει μεταφορά κονδυλίων από τα διευθυντικά ταμεία στο ΕΦΣΥ. Αυτή ήταν μια επιθυμία πολλών. Οι αρμοδιότητες ε, της Επιτροπής σχετικά με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων διατηρούνται. Επίσης, κάποια άλλα σημεία στα οποία συμφωνήσαμε ήταν ε, ότι αφορά τις επιδόσεις, τι, ε, πώς θα μετρούνται οι επιδόσεις, ποιες θα είναι οι παράμετροι. Μετά, ε, κόστος βασισμένο σε αποτελέσματα και σε αυτό συμφωνήσαμε, εσωτερικές ε, διαδικασίες, εδώ το Συμβούλιο θέλει να γίνουν ορισμένες αλλαγές, όμως σε αυτό το οικονομικό έτος έχουν χαθεί ορισμένοι πόροι και γι' αυτό θεωρώ πως πρέπει να ε, αντισταθούμε έτσι ώστε να μην χαθούν ακόμα περισσότεροι. Μετά, ευελιξία, αποθεματικό ταμείο έκτακτης ανάγκης. Εδώ πρέπει να περιμένουμε την έγκριση του Συμβουλίου. Χρειάζεται ακόμα δουλειά ε, έτσι ώστε να τροποποιηθεί ο ε, κανονικοσμός για το σε δημοσιονομικό πλαίσιο. Επίσης, ε, συζητήσαμε την ε, νέα διαδικασία έγκρισης, τις νέες μορφές συγχρηματοδότησης στα πλαίσια του ΕΦΣΥ. Εδώ προσπαθήσαμε να απλουστεύσουμε τα πράγματα. Στο πλαίσιο αυτό καταφέραμε να συμφωνήσουμε να συμπεριλαμβάνονται στον ε, κανονισμό πλαίσιο για το ΕΦΣΥ ορισμένα στοιχεία από αυτά που επιθυμούσαμε. Μετά ε, ζητήσαμε επιτάχυνση της διαδικασίας απαλλαγής και αυτό οδήγησε σε μια κοινή δήλωση που αναφέρει την κοινή επιθυμία επιτάχυνσης της διαδικασίας αυτής σε σχέση με τη σημερινή διαδικασία νησιν 2. Τώρα, η σχετική έκθεση έχει ήδη ε, προγραμματιστεί για προσυζήτηση και ψηφοφορία τον Ιούνιο, έτσι ώστε η απαλλαγή να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Αυτά λοιπόν σύντομα από μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω... Να ευχαριστήσω όλους και την ε, κυρία Γιάλα Σέντερ και όλους τους συναδέλφους που ε, εργάστηκαν σε αυτό το πολύ δύσκολο θέμα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τη Γραμματεία εδώ της Επιτροπής, όλους όσοι λοιπόν συνεργάστηκαν και προσπάθησαν πάρα πολύ. Θα δώσω όμως τώρα το λόγο στον συνάδελφο Ρίτσαρτ. Um, <clears throat> thank you, Chairman. Well, I too have few words of Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να πω κάποιες ευχαριστίες και να πω ότι η διαδικασία ήταν μακρά και χαίρομαι που αναφέρω ότι ολοκληρώσαμε τη διαδικασία και ήθελα να σχολιάσω ότι η εκπόνηση αυτού του κανονισμού πάντα είναι μια άσκηση ισορροπίας. Ευθύ εξ αρχή, ε, όλες οι πλευρές προσέγγισαν το θέμα με στόχο να υπάρξει απλοποίηση του συστήματο. Ε, Ιδίω απλοποίηση για τους χρήστε μέσω μείωσης γραφειοκρατίας. Αφετέρου βέβαια θα πρέπει να γνωρίζουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι ε, ε, οι διαδικασίες ελέγχου του συστήματος είναι αρκετά εύρωστες για να ελέγχουν ε, την κατάχρηση πόρων και επίσης θέλουμε να δούμε και αν μπορούμε να έχουμε προπολογισμό βάσει επιδόσεων. Είναι σαφές ότι για το μέλλον θα υπάρχει σπάνιδα πόρων, επομένως η διαδικασία λήψη αποφάσεων σίγουρα θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο στα αποτελέσματα και να υπάρχει και καλύτερη ενημέρωση. Με χαρά λοιπόν αναφέρω ότι μέσω αυτού του κανονισμού έγιναν τα πρώτα βήματα προς αυτή τη διαδικασία. Ε, είναι μακρύς ο δρόμος βεβαίως, αλλά νομίζω ότι αυτά τα οποία καταφέραμε είναι να έχουμε μία σειρά από κανονισμούς τα οποία θα δημιουργήσουν μια νέα νοοτροπία ε, κατάρτισης προπολογισμού βάσει επιδόσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θα ήθελα περισσότερη απλοποίηση, αλλά πρέπει να παραδεχτούμε ότι ο προπολογισμό βάσει επιδόσεων σημαίνει αυτονόητα περισσότερε διαδικασίε ελέγχου και όχι λιγότερε διαδικασίε ελέγχου. Και νομίζω ότι βάσει αυτού καταφέραμε να έχουμε ένα ισορροπημένο αποτέλεσμα. Η πρόοδο ανέφερα κάποια θέματα, απλοποίησαμε τη διαδικασία για την, ε, τα, τις επιδόσεις, ε, δώσαμε μεγαλύτερη έμφαση στις πληρωμές βάσει ε, αποτελεσμάτων και αναλογικότητα στα συστήματα ελέγχου και παρακολούθησης. Νομίζω ότι η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου παρέμεινε, ενισχύσαμε ίσως και τη θέση μας όσον αφορά τον έλεγχο του προπολογισμού έχουμε μία αρχή μη κέρδους ε, για τις ενισχύσεις και καταφέραμε να εξετάσουμε και όλα αυτά τα καταπληστευματικά ταμεία ε, και για το τι γίνεται με την ιστορική τους διαχείριση. Και πρέπει η Επιτροπή τώρα να κάνει αποτελεσματική χρήση αυτής της ρήτρας. Κατά την άποψή μου αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξει την οτροπία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι ε, ο Επίτροπος Έντεγκερ το εξετάζει το θέμα αυτό και θα ήθελα κυρία Πρόεδρε να ευχαριστήσω όλους εκείνους που συνεργάστηκαν. Θα πρέπει να αναφέρουμε και ε, την κυρία Σάιερ από την Προεδρία που κληρονόδότησε τη δουλειά και πρέπει λοιπόν να ευχαριστήσουμε και την Άντια Καλβίνο και την ομάδα της από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον πρόεδρο της Επιτροπής ε, ε, Προϋπολογισμών, τον κύριο Αρτουή, που πάντα ε, ήταν διαθέσιμος, τους σκιοδησηγητές, την Ινές κυρίως, και Μάσιμο να ευχαριστήσω και σα, κυρίω συγγνώμη, να ευχαριστήσω και εσά, κυρία Πρόεδρε, που ασχοληθήκατε με το θέμα αυτό, που κάνετε αξιοσημείωτη δουλειά και πραγματικά σα ευγνωμονούμε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι σπίτι. Είναι Σαγιάλα. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα απλώς για να το θυμόμαστε και γιατί όλες αυτές οι διαδικασίες έχουν ένα αντιφατικό στοιχείο. Δηλαδή, θέλουμε να έχουμε ε, καλύτερες προθεσμίες όσον αφορά τους ελέγχους, όπως πολύ σωστά είπε και η συγγήτρια, και να έχουμε έλεγχο νη συνένα και κατά την άποψή μου αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο αν υπάρχει ευρεία συνένεση μεταξύ όλων των οργάνων. Και όταν λέω όλα τα θεσμικά όργανα, περιλαμβάνω και τα κράτη-μέλη, διότι από εκεί απορρέει και μεγάλη σειρά των προβλημάτων, αλλά και των άλλων θεσμικών οργάνων που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα σε μικρότερο χρονικό διάστημα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να βελτιωθεί και η ποιότητα. Να πω ότι κάθε φορά που ξεκινάει η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού, εγώ ε, θα απαιτήσω ε, ο εισηγητής, ο εισηγητής να μας πούνε σε πόσους μήνες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Χρειάζεται ένα χρονοδιάγραμμα και για μας να το γνωρίζουμε και να ξέρουμε ότι δεν θα χάσουμε ένα κομμάτι τη ζωή μας σε αυτές τις ατέρμονες ε, συνεδριάσεις κάθε χρόνο για τέλειο τους μήνες. Ξεκινήσαμε με δύο εισηγητέ από την ε, Επιτροπή Προπολογισμών και την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, καθένα από διαφορετική πολιτική ομάδα, που μα έδινε όπω γίνεται ιστορικά πλειοψηφία και μετά από πολλού μήνε έγιναν τα σημαντικά βήματα ώστε να καταλήξει στα χέρια μια ομάδα. Γιατί ο κύριο Άσουορ τελικά ε, βρέθηκε και στο ΕΛΚ. Έχουμε ένα κανονισμό που μετά από μήνε ε, ε, καλή συντροφικιά θα μπορούσαμε να πούμε, μπορούμε να υποστηρίξουμε σε γενικές γραμμές, αλλά νομίζω ότι σε άλλη περίπτωση θα πρέπει να βελτιώσουμε και τη διαδικασία. Συγκεκριμένε προθεσμίες για να μην απελπιζόμαστε και να περνούμε μήνε εργασία, και να είμαστε βέβαιοι ότι ο πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνενεί για την όλη διαδικασία γιατί δεν θέλουμε να εξαπατήσουμε και τους υπολείπους, ε, τα υπόλοιπα μέλη του Κοινοβουλίου. Θέλω τουλάχιστον στο μέλλον να γίνει αυτό. Όσον αφορά το αποτέλεσμα δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο, συμφωνώ απόλυτα γιατί οι προσπάθειες ήταν τεράστιες. Να ευχαριστήσω και εγώ και τον κύριο Μα που αποσιάζει εδώ γιατί έχει προβλήματα με τις μεταφορές αλλά συνεργάστηκε μαζί μας, τη γραμματεία φυσικά της ομάδας μας που ασχολήθηκε και αυτή ώρες ολόκληρες ε, μαθαίνοντας με ποιο τρόπο μπορούν να διευκολύνουμε τους δικαιούχους ε, ε, να έχουν πιο εύκολες διαδικασίες, διότι εκεί έξω, ε, εγώ στο προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην περιφέρειά μου είδα ότι όλοι αυτοί που δικαιούνται κονδύλια είναι όλο ένα και πιο απογοητευμένοι, χρειάζεται όλο ένα και περισσότερη γραφειοκρατία, δικαιολογητικά, αποδεικτικά στοιχεία. Πρέπει κάποια στιγμή λοιπόν να προσπαθήσουμε ε, όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο εφαρμογής αυτή σε άλλους τομείς ε, και σε τοπικό επίπεδο, θα μπορέσουμε να περιορίσουμε αυτή την τεράστια ποσότητα ε, εγγράφων και τόσο περίπλοκων στοιχείων που τους ζητάμε. Ήταν μια διαδικασία απλοποίησης, να συγχαρώ και την ησυχήτρια για την τεράστια προσπάθεια που έκανε και που έδειξε και τη διάθεση να καταλάβει και να τη ρωτήσω, γιατί θα ήθελα να μπορέσουμε να το πούμε και φωναχτά δημοσίω, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσον αφορά τον έλεγχο των ε, αποκεντρωμένων υπηρεσιών και οργανισμών να μπορούν να, ε, για να διευκολύνουν και τη δουλειά του ελεγκτικού συνεδρίου αυτές οι έλεγχοι να γίνονται με ε, δημόσια κονδύλια και όσοι ασχολήθηκαν και με τη συνεργασία με το Συμβούλιο, άλλαζαν οι προεδρίες και κάθε προεδρία έπρεπε να μάθει από την αρχή τι συζητούσαμε και ήταν πολύ μεγάλες οι δυσκολίες. Πρόκειται λοιπόν για ένα γκάφι το οποίο πρέπει να ε, λύσουμε όταν βλέπουμε τι πρόβλημα υπάρχει με τις απαλλαγές των υπηρεσιών και οργανισμών και πόσο δύσκολο είναι να γίνει έλεγχος, πρέπει κάποια στιγμή να συμφωνήσουμε με το Συμβούλιο, να υπάρχουν επαρκείς πόροι, να υπάρχουν αρκετά κονδύλια ώστε να μπορεί να γίνονται δημοσίως αυτοί οι έλεγχοι και να είναι πλήρης ο έλεγχος και ε, να γίνεται από το ελεγκτικό συνέδριο. Να ευχαριστήσω τους πάντες, τη Γραμματεία της Επιτροπής, την ομάδα της κυρίας Καλβίνια και τον κύριο Ολιβιέ για την προσπάθεια που έκαναν προκειμένου να καταφέρουμε να έχουμε ένα αίσιο τέλος και να ευχαριστήσω και τους εισηγητές. Also, was das Thema Entlastung betrifft. Όσον αφορά και το θέμα των απαλλαγών, αν κατάλαβα καλά, θα πρέπει να δούμε τελικά πώς μπορούμε να συντομεύσουμε τις διαδικασίες, χωρίς βεβαίως να θέσουμε σε κίνδυνο την όλη διαδικασία και την αξιοπιστία σας. Πώς μπορούμε εκ των προτέρων να δούμε τις προθεσμίες, γιατί καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές ε, η όλη διαδικασία μπορεί να αποτύχει λόγω αυτού. Υπάρχουν, όπως ξέρετε, πάρα πολλά εμπόδια που τίθενται λόγω υποχρεώσεων των κρατών μελών, ημερομηνίες οι οποίες ε, δυσκολεύουν το ένα ή το άλλο κράτος μέλος. Σήμερα βλέπουμε ότι οι διαδικασίες αυτές επιμηκύνονται και οι διαδικασίες των απαλλαγών καθυστερούν υπερβολικά και όσον αφορά τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και οργανισμούς δεν μπορέσαμε να βρούμε εδώ κοινά σημεία και όσον αφορά αυτό που αναφέρατε για την διεξαγωγή όλων αυτών των επαληθεύσεων και ελέγχων από δημόσια κονδύλια, με χρηματοδότηση δημόσιων κονδύλιων, αλλά και για τον συντονισμό και για κάποιες κοινέ Σας Ευχαριστώ και εγώ πολύ όλους όσους συνεισφέρετε σε αυτή τη ε, δουλειά. Thank you, Chair. It's my turn to... Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και τον κύριο Άσφορτ και την κυρία Αγιάλα για τα πολύ θετικά σας λόγια όλοι. Χαίρομαστε ιδιαίτερα που μπορέσαμε να προχωρήσουμε στο έργο. Αυτό ήταν ε, πολύ σημαντικό για την Επιτροπή να υπάρξει ένα σταθερό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορέσουμε να δουλέψουμε και να προετοιμάσουμε τους ε, νέους άξονες, τις νέες κατευθυντήριες γραμμές για το δημοσιονομικό πλαίσιο, λοιπόν, είμαστε ευτυχείς που έχει διασφαλιστεί το πλαίσιο αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ όλους. Θα θέλαμε εδώ να υπογραμμίσουμε τη σημαντικότατη, αν θέλετε, αυτή ε, διαδικασία η οποία θα θέλαμε το συντομότερο δυνατόν να εγκριθεί. Ελπίζουμε, ελπίζουμε τον Ιούλιο φέτος. Ναι, αυτό έχουμε προλέψει. Μία προϋπόθεση όμως σημαντική είναι να έχουμε ένα κείμενο το οποίο μπορεί να ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Δεν βλέπω κάποιον άλλο που θέλει να πάρει το λόγο, οπότε περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, το ψήφισμα. Δύο λεπτά να διαβάσω το σωστό, πολιτική της ευρωπαϊκής πολιτικής που αφορά το θέμα της ε, ακυρεότητας της και ειδικότερα ο διορισμός του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το κείμενο το έχετε, όπως το έχουμε υποβάλει. Σκοπός αυτής της ε, αν θέλετε, διαδικασίας είναι να ανακληθεί η διαδικασία και να ακολουθηθεί μια διαδικασία να ακολουθηθεί μια άλλη διαδικασία. Καταλαβαίνετε ότι τα στοιχεία περιγράφονται εδώ και θα πρέπει να περιγράφονται με αντικειμενικό τρόπο το θέμα της σταδιοδρομίας, σταδιοδρομίας και των προηγούμενων γενικών γραμματέων, η διαδικασία διορισμού, η αξιολόγηση, αυτό που αν θέλετε προσπαθήσαμε εδώ να κάνουμε είναι να κοιτάξουμε λιγάκι και το μέλλον. Δηλαδή το θέμα της νομικής βάσης. Όσον αφορά αυτό το κομμάτι, εγώ βεβαίως ε, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Το θέμα, αν θέλετε, του πώς μπορούμε να απο, αποπέμψουμε έναν γενικό γραμματέα, είναι κάτι για το οποίο νομίζω δεν υπάρχει προηγούμενο. Είναι η συζήτηση γύρω από την νομική βάση είναι κάτι που βεβαίως ε, είναι πολύ ενδιαφέρουσα, αλλά μέχρι τώρα βασιζόμαστε στον κανονισμό του προσωπικού και αυτό είναι η βάση. 29 είναι οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί. Κοιτάξτε, εγώ ήμουνα στη Λετωνία την προηγούμενη εβδομάδα και στη Λιθουανία με το θέμα αυτό. Λοιπόν, δεν μπόρεσα να ασχοληθώ. Ο κατάλογος για τις ψηφοφορίες Κοιτάξτε, εγώ για ποιο λόγο απορρίπτω όλες τις ε, τροπολογίες και γιατί σας προτείνω να κάνετε το ίδιο κι εσείς. Πρώτον, πιστεύω ότι το κείμενό μας συμπεριλαμβάνει όλα τα σημαντικά σημεία και πιστεύω ότι η συμβουλή που λάβαμε είναι εξαιρετικά καλή δεν πιστεύω ότι πρέπει να οξύνουμε περισσότερο τα πράγματα. Το κείμενο συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία, όλα τα σημεία εκεί που δεν τηρήθηκε σωστά η διαδικασία. Ε, όσον αφορά, αν θέλετε, το κείμενο, δεν θέλω να γίνει ούτε πιο οξύ, ούτε πιο αδύναμο σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, πιστεύω ότι εδώ δεν θα πρέπει βεβαίως ε, να αποφασίσω μόνη μου. Υπάρχουν οι εισηγητές, υπάρχουν οι συντονιστές. Εγώ βεβαίως έχω μία, μία ψήφο. Επαναλαμβάνω το θέμα της νομικής βάσης, επαναλαμβάνω και το θέμα του άρθρου 50 του κανονισμού του προσωπικού που είναι, αν θέλετε, αυτό στο οποίο πρέπει και μπορούμε να βασιστούμε. Με 15.000 ευρώ το μήνα καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν θα αφήσει μια τέτοια θέση για να φύγει, αλλά οι μέχρι τώρα ενσωματωμένες αλλαγές και τροποποίησεις που προτείνατε έχουν σαφώς βελτιώσει το κείμενο, Γι' αυτό και θεωρώ ότι τις υπόλοιπες τροπολογίες ε, δεν θα πρέπει να τις δεχτούμε. Ακούσαμε και την ε, νομική υπηρεσία, η κυρία Μοντεμπέλο. Είναι παρούσα από την ε, νομική υπηρεσία, δεν την είχα δει, ζητώ συγγνώμη, αν έχετε ερωτήσεις σαφώς και είναι εδώ στη διάθεσή μας. Υπάρχει και το δεύτερο ερωτηματολόγιο Μπορείτε να τοποθετηθείτε επ' αυτού. Εάν θέλετε να πάρετε το λόγο βεβαίως για αυτό το θέμα, σας το δίνω αμέσω. Merci, merci Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Τι να σας πω. Η Επιτροπή έχει υποβάλει κάποιες προσπάθειες, θα έλεγα, δικαιολόγησης, αιτιολόγησης, δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπήρξε δημοσίευση, ο συγκεκριμένος ε, υπάλληλος ε, μένει, παραμένει με τη θέση του. Για ποιο λόγο. Πρώτον, εμπιστοσύνη μεταξύ του δημάσου Υπαλλήλου και του Προέδρου της Επιτροπής, η συνέχεια της ε, παροχής υπηρεσιών, οι εξαιρετικές αυτές προϋποθέσεις που ουσιαστικά αφορούν και την εξαιρετική περίπτωση λόγω Brexit. Αυτό δεν μπορεί η νομική υπηρεσία να το αξιολογήσει. Αυτό που θα ήθελα εδώ να πω όσον αφορά την αντικειμενική μας γνωμοδότηση, όπως σας την υποβάλαμε, βασιστήκαμε στην ομολογία Τούρκο Εκεί υπάρχει ίσως μια διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά τη νομική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω και επιμένουμε σε αυτό ότι για αυτές τις θέσεις η δημοσίευση είναι η ισχύουσα πρακτική και μια εξαιρετική, αν θέλετε, περίπτωση όπως αυτή που προτείνει εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να παραμείνει δηλαδή η θέση ε, είναι κάτι το πολύ εξαιρετικό. Εδώ λοιπόν θα πρέπει, όπως είπατε και εσείς, να ισχύσει ο κανονισμός και ενδεχομένως θα πρέπει, αν ο κανονισμός αυτός εμπεριέχει αδυναμίες ή κενά, να το λάβουμε υπόψη μας για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Φυσικά και θα λάβουμε υπόψη το ερωτηματολόγιο, που είναι πάρα πολύ μεγάλο. Λοιπόν, προτείνω ε, να δούμε αν θέλει κάποιος το λόγο. Ε, Ίνες, Ίνες, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ για την προσπάθεια που έγινε, αν και πρέπει να πω ότι θα μπορούσε ίσως να ήταν πιο λογικό να κάνουμε ένα πιο σύντομο ε, ψήφισμα και να μπορέσουν έτσι οι βουλευτές ε, να υποβάλουν τροπολογίες. Γιατί τώρα να λέτε ότι δεν θα γίνουν δεκτές οι τροπολογίες, ε, καταρχήν δεν είναι αποδεκτό για το Κοινοβούλιο. Δεύτερον, μόλις είπες και ψάχναμε να βρούμε και με ποιο τρόπο ε, μπορούμε να δούμε τη βάση για το Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με εκπλήσει το γεγονός ότι δεν έχουμε καν βάση. Και νομίζω ότι και ο κύριος Έτιγκερ έκανε μια προσπάθεια την οποία αναγνωρίζω, δηλαδή πρόσφερε τη δυνατότητα να συζητήσει με το Κοινοβούλιο για να δει πιθανή αναθεώρηση των κανόνων, διότι αυτό το οποίο κατέστησε σαφές είναι ότι ναι, μεν το επέτρεπε οριακά ο κανονισμός, ε, ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόστηκε ο κανόνας ε, ε, βάσει των εξηγήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μας οδήγησε στην κατάσταση που βρισκόμαστε σήμερα, που δεν είναι καλή ούτε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτε για κανένα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Επομένως θεωρώ ότι πρέπει με σαφή τρόπο να πούμε ότι πρέπει να γίνει αναθεώρηση των κανόνων. Δεν μπορεί να παρετήσουμε και ένα γενικό γραμματέα, ο οποίο μπορεί να κάνει το οτιδήποτε. Δεν αναφέρομαι στον κύριο Σελμάγερ, αναφέρομαι γενικότερα. Δεν αναφέρομαι σε κανέναν, μην με παρεξηγήσετε, οποιονδήποτε γενικό γραμματέα, ο οποίο θα μπορούσε στο μέλλον ή θα έχει δημιουργήσει προβλήματα και στο παρελθόν, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει τρόπος να υπάρχει και μια πρόταση μομφής εναντίον του. Ε, πρέπει λοιπόν να πούμε σαφέστατα ότι οι κανόνες έχουν προβλήματα. Ε, πρώτα λοιπόν θα πρέπει να πούμε κάπως ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε τους κανόνες διότι ε, η ιδιότητα του Γενικού Γραμματέα που είναι ε, ουσιαστικά ε, ο επικεφαλής όλης της διοικητικής διαδικασίας και κάθε πέντε χρόνια που αλλάζουν ε, τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, δεν γίνεται να αλλάζει, αλλά πρέπει να βρούμε τρόπο να τα κάνουμε, να αλλάξει ο κανονισμός. Αν δεν γίνει η αλλαγή τώρα θα γίνουν χειρότερο και όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε άλλα θεσμικά όργανα που γνωρίζουμε όλοι τι συμβαίνει. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό να ζητήσει αναθεώρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι ο κύριος Έτιγκερ μας έδωσε ουσιαστικά τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε μια τέτοια διαδικασία. Δεύτερον, εγώ πιστεύω και το είπαμε και από την ομάδα μα, αν και θα πρέπει να γίνει συζήτηση και στο Κοινοβούλιο, ε, μάλλον η συζήτηση για το Κοινοβούλιο, για την Ολομέλεια αυτή την εβδομάδα, δεν υπάρχει κανένα στοιχείο άμεσης σταθερότητα, γιατί αυτή τη στιγμή συζητούμε το Brexit, θα ξεκινήσει η συζήτηση για τον προπολογισμό. Ε, έχουμε και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα φρικτά πράγματα, αυτά τα οποία συμβαίνουν και με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις απειλές για το διεθνές εμπόριο ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν θεωρώ ότι είναι στιγμή να ανοίξουμε το κουτί της Πανδώρας χωρίς να ξέρουμε και προς τα που οδεύουμε, γιατί τα κάναμε αυτά στο παρελθόν και ξέρουμε και που καταλήξαμε. Θα πρέπει δηλαδή ως προς την ευθύνη μας, ε, επειδή είναι και έτσι όπως είναι η κατάσταση και τη σχέση έχει δημιουργηθεί μεταξύ του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του νέου Γενικού Γραμματέα, ε, θεωρώ ίσως ότι αυτή τη στιγμή και με τους παρόντες κανόνες που είναι σαφές ότι δεν είναι καλή, δεν πρέπει να κάνουμε κάτι παραπάνω. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν οι κανόνες, σίγουρα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Πρέπει δηλαδή να πούμε ότι η Νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να συνεχίσει ως συνήθως. Αν υπάρχουν νέους, νέοι κανόνες θα πρέπει να αναθεωρηθούν οι αποφάσεις. Δεν έχω τίποτα κατά του κ. Σελμάγερ ως ατόμου, δεν το γνωρίζω κιόλας αλλά σίγουρα θεωρώ ότι η θέση ε, προκειμένου να είναι πιο ισχυρή και η Κοινή Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να μην είναι αποδυναμωμένη, είναι να αναθεωρηθεί απόφαση. Αν θέλει να είναι υποψήφιος ο κύριος Ελμάγερ, ε, να είναι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αλλά ε, όσον αφορά τώρα το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας οφείλει τη δυνατότητα να έχουμε γνώμη. Δεν με αναφέρουμε σε δυνατότητα ε, βέτο, γιατί εγώ συμφωνώ για την ανεξαρτησία των θεσμικών οργάνων και η διοργανική συμφωνία θα πρέπει να ε, θεμελιώνει και ένα κατάλληλο διάλογο για να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Αυτή τη στιγμή είμαστε παραμονή ε, του να δώσουμε τη σύμφωνη γνώμη μας για τον Γενικό Γραμματέα της Όλαφ και νομίζω ότι όσον αφορά τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα όσα συνέβησαν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας οφείλει να αναθεωρήσουμε τους κανόνες, να ξαναδούμε τα πράγματα όταν θα τελειώσει η θητεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το Κοινοβούλιο πρέπει να έχει λόγο. Νομίζω αυτά τα τρία πράγματα θα πρέπει να βρίσκονται σε μελλοντική συμφωνία για να μην ξανασυμβούνται αυτά τα οποία συνέβησαν. Also, Λοιπόν, αν διαβάσει κανείς το κείμενο, τότε βλέπουμε ότι φυσικά και υπάρχει μέσα αυτό το θέμα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ως συμβιβασμό. Αυτές οι επίμαχες τροπολογίες όπου αναφέρεται η σχέση ανάμεσα σε, αυτήν, ε, την, ε, σε αυτόν τον ξαφνικό διορισμό και στην ε, φυσιολογική εξέλιξη μιας ε, σταδιοδρομίας, θα μπορούσαμε να τις κοιτάξουμε. Νομίζω πως υπάρχουν ορισμένες ε, πολύ σωστές απορίες, πολύ σωστές αντιρρήσεις που έχετε, που έχουν οδηγήσει σε αυτές τις ε, πολύ λογικές και αναμενόμενες αντιδράσεις με όλη αυτή την ιστορία. Πιστεύω πως το ψήφισμα περιέχει σημεία τα οποία ε, ασκούν φυσικά δερμία κριτική, η οποία όμως είναι πολύ δικαιολογημένη. Ο κύριος Εντεγιόν έχει το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να σας συγχαρώ για την πολύ λεπτομερή ανάλυση αυτού του θέματος. Πιστεύω πως έχετε ταπανίσει πάρα πολύ χρόνο και κόπο πάνω σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό λοιπόν και από μένα δεν ήρθαν πολλές τροπολογίες. Όμως, το θέμα εδώ δεν είναι το πώς ε, θα διαπιστώσουμε τη λειτουργία ε, του κανονισμού σχετικά με το διορισμό των ανώτερων υπαλλήλων. Το θέμα είναι να ε, κοιτάξουμε τη δημόσια εικόνα μας, η οποία πλήττεται από αυτό. Και όπως ακριβώς ασκούμε έλεγχο στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς, έτσι πρέπει να γίνει και στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ε, το θέμα εδώ όχι το τι έγινε και πώς ε, εφαρμόστηκε ο κανονισμός. Αλλά το θέμα έχει ως εξή, Όταν πέφτει το κάποιο από το πουθενά με αυτόν τον τρόπο, ε, τότε γίνονται θέματα διαφάνειας. Και ιδιαίτερα στην περίπτωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που βρίσκεται συνέχεια στα μέσα ενημέρωσης, ε, που είναι η δημόσια εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και εμείς, όπως και το Κοινοβούλιο. Και φυσικά πρέπει να λάβουμε μέτρα έτσι ώστε να μην λάβει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις το θέμα αυτό. Έχουμε διαβάσει πάρα πολλές ε, σχετικές αναφορές και αναλύσεις ε, για το θέμα. Το έχουμε συζητήσει ήδη πάρα πολύ. Σίγουρα ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έπρεπε να είναι ενήμερος για όλα αυτά. Δεν γίνεται αλλιώ. Τώρα. Μετά. Κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση. Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, χρειάζεται προσοχή σχετικά με το ότι αυτές οι διαδικασίες μπορεί και να καταλήξουν ενώπιον του δικαστηρίου. Πρέπει να διαβάσουμε με μεγάλη ε, προσοχή το τι έχει συμβεί. Υπήρχε, λέει, ένα ε, σχέδιο Β, το οποίο ήταν ήδη καταρτισμένο σύμφωνα με ε, το οποίο είχαν προβλεφθεί διάφορες ενέργειες σε περίπτωση που υπήρχαν προβλήματα. Και σίγουρα αυτά θα έπρεπε να τα ξέρουν οι πρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς χρειαζόμαστε ένα φεδρικό σχέδιο, βέβαια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Διότι είναι και θέμα εμπιστοσύνης. Το σώμα των επιτρόπων αποτελείται από άτομα τα οποία ανήκουν σε διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και πρέπει να υπάρχει γενικότερη ομοφωνία και νομίζω πως εδώ είναι το ζητούμενο. Πρέπει να προσέξουμε το τρόπο με τον οποίο έγινε η διαδικασία και το πόσο μονομερής ήταν η, απόφαση ή όχι. Και σίγουρα πρέπει να δείξουμε την αλληλεγγύη μας προς ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και τρίτον, τα μέσα ενημέρωσης. Ο τύπος, δημοσιογράφοι, να σας πω ότι ποτέ δεν έχει ξανατύχει να ακούσω σε συνεντεύξεις τύπου, όταν αναφέρεται τέτοιο θέμα, να αποσιωπάτε τόσο γρήγορα. Εδώ, στο ψήφισμα υπάρχουν ορισμένες τροπολογίες, οι οποίες όχι μόνο αναφέρουν το θέμα αυτό, αλλά περνάνε και σε ένα στάδιο παραπέρα. Δεν είμαι 100% σίγουρος για το κατά πόσο πρέπει να βρίσκονται σε αυτό το ψήφισμα αυτές οι τροπολογίες. Αλλά όπου γίνεται αναφορά στο ότι ο Γενικός Γραμματέας θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αρνηθεί τον διορισμό του, είναι κάτι που πρέπει να δούμε. Ίσως αυτό είναι και προς το συμφέρον όλων, ιδιαίτερα εν ώψη των διαπραγματεύσεων για το Brexit. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή όταν ο πρόεδρος της ε, Κομισιόν εξαρτάται τόσο πολύ από τον, ε, από τον Γενικό Γραμματέα, τότε ε, δημιουργούνται προβλήματα. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια εξάρτηση ανάμεσα στον πρόεδρο της Κομισιόν και στο Γενικό της Γραμματέα. Αυτό είναι πολύ νευραλγικό θέμα. Αυτό και άλλα πολλά είναι πολύ σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να συζητήσουμε πρωτού ψηφιστεί στην Ολομέλεια το παρόν ψήφισμα. Και όπως είπα χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Εμείς ως Επιτροπή Ελέγχου του προπολογισμού πρέπει να προσέξουμε και για να μην αμαυρωθεί η δημόσια εικόνα της Ευρωπαϊκή Ένωσης. Να αποφύγουμε οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση της κατάστασης να πάρουμε το θέμα αυτό στα σοβαρά και να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι οι πράξεις έχουν και συνέπειες. Και όταν αυτές οι συνέπειες οδηγούν σε άσχημη εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ευχαριστώ, κύριος Κυρπράντη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόταση αυτή ψηφίσματος. Θα συμφωνήσω και εγώ με του συναδέλφους ότι είναι αρκετά έντονα τα λόγια του ψηφίσματο και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Ωστόσο, η δική μου πολιτική ομάδα θεωρεί πως χρειάζονται ορισμένε βελτιώσει Για τον λόγο αυτό, υποβάλαμε ορισμένες λίγες τροπολογίες, ακριβώς διότι πιστεύουμε πως ε, είναι πολύ σημαντικό να γίνουν κάποιες βελτιώσεις. Τώρα, Ορισμένα σχόλια από μένα. Εάν υπάρχει ένα θεσμικό όργανο που μπορεί να ελέγξει δημοκρατικά την Κομισιόν, είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν υπάρχουν ε, θέματα όπως πολιτικοί διορισμοί εντός ενός θεσμικού οργάνου, νομίζω πως ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το καθήλυν αρμόδιο για να ασκήσει έλεγχο. Και δεν συμφωνώ ε, με όσους λένε πως αυτό είναι θέμα της Κομισιόν και δεν έχει δουλειά το Κοινοβούλιο εκεί. Τώρα, εάν και κατά πόσο ε, όλο αυτό το σκηνικό οδηγεί σε ε, επιδείνωση της εικόνας της Κομισιόν ή όχι. Αυτό πιστεύω πως δεν έχει τόσο σημασία. Η ίδια η Κομισιόν πρέπει να κληθεί να απαντήσει και να αναλογιστεί το, σχετικά με το πώς χρησιμοποίησε τον εσωτερικό της κανονισμό. Και τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, συνέντευξη τύπου της Κομισιόν, να πω πως εντάξει δεν ήταν και ιδανικό, δεν ήταν και υπόδειγμα επικοινωνίας αυτή η συνέντευξη τύπου. Τι περιμένω περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραδεχτεί ότι η διαδικασία που ακολούθησε δεν ήταν ιδανική. Το κάθε άλλο. Μας ε, απέστειλε ένα πάκο απαντήσεις. Ο κύριος Σέτινιερ ήταν άφαντος, απέφυγε να απαντήσει και στο δεύτερο ε, κομμάτι των γραπτών απαντήσεων που μας έστειλε η Επιτροπή δεν είδα καμία παραδοχή πουθενά για το ε, πόσο κατάλληλη ή πόσο κατάλληλη ήταν η διαδικασία που ακολουθήθηκε. Και αυτό είναι το πρόβλημα που έχω. Μπορούμε φυσικά να ασκήσουμε δρυμύτατη κριτική, όμως χρειάζεται πρώτα η ίδια η Κομισιόν να ασκησουμε την κριτικη ομως χρειαζεται πρωτα η ιδια η κομισιον να παραδεχτει ε, το λάθος της. Μετά το κατά πόσο ήταν πολιτικός ο διορισμός. Ε, το ότι ο Γενικός Γραμματέας αναλαμβάνει καθήκοντα τα οποία θα επεκταθούν και μετά το τέλος της θητείας αυτής της Επιτροπής. Δεν είμαι καθόλου υπέρ της πολιτικοποίησης της θέσης του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θεωρώ πως υπάρχουν πολιτικά επιτελεία για όλους τους επιτρόπους και πως οι υπόλοιποι υπάλληλοι πρέπει να είναι όσο το δυνατόν ε, πιο ουδέτεροι. Αυτό συμπεριλαμβάνει και τον Γενικό Γραμματέα. Τώρα, εάν ο νέος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αντιμετωπίσει ιδιαίτερε δυσκολίες στη συνεργασία του με τον Γενικό Γραμματέα της ε, Κομισιόν, τότε αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για να δημιουργηθεί μια διαδικασία εξέτασης της πιθανής αποπομπής του Γενικού Γραμματέα. Όμως ε, πιστεύω πως ε, αυτό που γίνεται τώρα δεν είναι σωστό. Δεν είναι ο σωστός δρόμος. Αν θυμάστε καλά, ο κύριος ε, Ιταλιάνερ, ο προηγούμενος Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είχε έναν αμφιλεγόμενο ρόλο. Δεν νομίζω πως πολλοί γνωρίζουν το ρόλο που διαδραμάτισε ήταν ουδέτερος θα μπορούσε να το πει κανείς αφανής θα μπορούσε να το πουν άλλοι ιδιαίτερα σε σχέση με την Κάθιν ε, Τέι, την πρωτοκάτοχό του. Τώρα, εδώ στην Επιτροπή, πιστεύω πως ε, θα πρέπει να ψηφίσουμε την επόμενη εβδομάδα τις τροπολογίες που υποβλήθηκαν για το ψήφισμα, να δούμε τι θα γίνει στην Ολομέλεια. Πιστεύω όμως ότι ο πρόεδρος Γιούγκερ, ο οποίος είναι ο καθήλ αρμόδιος για αυτό το θέμα, θα πρέπει να σταθεί υπόλογος εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια. Εγώ θα ήμουν υπέρ μετά τη Δευτέρα το βράδυ, μετά την ψηφοφορία της Επιτροπής μας για το ψήφισμα αυτό, να γίνει μια συζήτηση με τον πρόεδρο Γιούγκερ παρόντα έτσι ώστε να συζητήσουμε το θέμα. και να δώσουμε στον πρόεδρο της Κομισιόν τη δυνατότητα να παραδεχτεί δημόσια ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν ήταν ιδανική. Κύριο κύριος Ευχαριστώ. Εγώ συμφωνώ μαζί σας, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά παθιασμένοι και εμπαθείς, να κοιτάξουμε την ουσία και να δείξουμε σαφώς υπευθυνότητα, γιατί το θέμα το απαιτεί. Κυρία Πρόεδρε, και προς εσάς και προς τους συναδέλφους θέλω να πω ότι στο σχέδιο ψηφίσματος αυτού υπάρχει η παραγραφός 18 ε, που αναφέρει ρητά ότι το Κοινοβούλιο αναφέρει αυτήν την διαδικασία διορισμού δύο φάσεων η οποία μοιάζει με πραξικοπηματική ενέργεια και είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά κάνει μία διασταλτική ερμηνεία του κανονισμού. Και πραγματικά από αυτό το κείμενο θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα μαθήματα που πρέπει να μάθουμε. Πέραν των μαθημάτων, κυρία Πρόεδρε, μήπως χρειάζεται και κάποια ενέργεια. Δεν απαιτείται από μας κάποια ενέργεια, κάποια δράση. Αυτή η δήλωση ουσιαστικά δεν μπορεί απλώς να γίνει και να μείνει χωρίς να ακολουθηθεί από καμία αποδηλήτως ενέργεια. Κυρία Πρόεδρε, αναφερθήκατε και στις τροπολογίες που έχει υποβάλει η συνάδελφος η Νέα Ουσιαστικά με αυτές τις ε, τροπολογίες ζητάμε από την Επιτροπή να μας υποβάλει το ταχύτερο δυνατόν, χωρίς καθυστερήσεις, την τελική της ε, πρόταση για αυτή την υπόθεση. Και δεν ξέρω. Εγώ σκεφτόμουν αυτή την τροπολογία, όχι κάποια άλλη. Εσείς κάποια άλλη θα θέλατε φαίνεται να δεχτείτε. Η 116 σε αυτή αναφέρομαι και πιστεύω ότι είναι ορθή αυτή η τροπολογία. Ουσιαστικά ρωτάει από την Επιτροπή τι προτίθεται να κάνει, ποια είναι η απαραίτητη ενέργεια και δράση που πρέπει να υιοθετηθεί. Γιατί λάβαμε από την Επιτροπή δεκάδες σελίδες ε, αιτιολογήσεων και μετά από ώρες ακροάσεων και συζήτησης δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το θέμα. Δεν έχω την εντύπωση δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει συνειδητοποιήσει ότι κάτι δεν πήγε καλά. Μα είναι δυνατόν. Αναρωτιέμαι ματικά πού βρίσκεται αυτή η Επιτροπή, σε ποιο πλανήτη. Ο προηγούμενος ομιλητής αναφέρθηκε στην μη πολιτικοποίηση της θέσης του Γενικού Γραμματέα. Αυτό είναι πολύ ορθό. Βρισκόμαστε όμως σε μια πάρα πολύ δυστυχή θέση και διαπιστώνουμε ότι έχει πολιτικοποιηθεί. Και αυτό εξαιτίας της παρούσας ε, περίπτωσης και διαδικασίας. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξαναδεί τα πράγματα, ότι πρόκειται για ένα πλέον πολιτικό θέμα και να μην απορρίψει την περίπτωση από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το ισχυρό αίτημα από μέρους μας, αυτή η πολιτικοποίηση της θέσης του Γενικού Γραμματέα να αντιμετωπιστεί με έναν τρόπο που δεν είναι αυτός που αντιμετωπίζεται αυτή τη στιγμή από την Επιτροπή. Κυρία Πρόεδρε, Σήμερα εδώ σε αυτή τη συνεδρία εξετάζουμε το ψήφισμα που προτείνεται κύριε Πρόεδρε και είναι μια πολύ σημαντική συνεδρίαση γιατί ουσιαστικά σήμερα καθορίζουμε ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πέρα λοιπόν ε, του ότι ζητάμε μια συζήτηση στην Ολομέλεια και ψηφοφορία υπάρχει και το αίτημα εμείς η Επιτροπή Ελέγχου του προπολογισμού, να παίξουμε τον ρόλο μας. Το ρόλο που εξάλλου πάντα παίζουμε. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για το κείμενο που μας υποβάλλετε. Όπως υπενθύμισε όμως τώρα μόλις ο συνάδελφος Κυπράντη, σε κάθε περίπτωση εμείς που θέλουμε και το επαναλαμβάνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παίξει έναν ελεγκτικό ρόλο εναντί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να βελτιώσουμε τις δυνατότητες που έχουμε. Διότι όντως άνοιξε το κουτί της Πανδώρας από το ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας. Και αυτό γιατί υπάρχουν ε, κενά στην διαδικασία που ακολούθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό το έχουμε διαπιστώσει, το έχουμε δει και στις 165 σελίδες απάντησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και όταν έγινε η ακρόαση 27 Μαρτίου του Επιτρόπου Έτιγκερ ο κύριος Έτιγκερ μας είπε ότι ο κύριος Ελμάιερ συμμετείχε στην ε, προετοιμασία αυτών των αποφάσεων. Αυτό είναι κατάφορη παραβίαση του άρθρου 11 του κανονισμού του προσωπικού. Βλέπετε λοιπόν ότι όλα αυτά τα στοιχεία είναι πολιτικά και έχουν ανοίξει το κουτί της Πανδάρος. Και όπως είπα και ενώπιον του Επιτρόπου Έτιγκερ, Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε εξάλλου και χτες με τα αποτελέσματα των εκλογών στην Ουγγαρία. Βλέπετε ότι το αντιευρωπαϊκό κίνημα διαρκώς ενισχύεται από το 2014 μέχρι σήμερα στα κράτη-μέλη. Θα πρέπει λοιπόν το ψήφισμά μας να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο να συνειδητοποιήσουν ότι αυτό το κουτί της Πανδώρας πρέπει να κλείσει. Πώς θα κλείσει το κουτί της Πανδώρας. Μόνο εάν βρούμε μια λύση που θα καθησυχάσει και θα ηρεμήσει τα πράγματα. Εδώ και δύο μήνες η διαδικασία αυτή διαρκώς οξύνεται. Εμείς λοιπόν πρέπει να υποβάλουμε ένα δυνατό κείμενο, ένα ισχυρό κείμενο που να δίνει απαντήσεις και να βοηθάει στο να κλείσει το κουτί της Πανδώρας. Πρέπει να ενισχύσουμε την αξιοπιστία των ευρωπαϊκών θεσμών. Δυστυχώς, με την υπόθεση Σελμάιερ, η αξιοπιστία μας έχει υποστεί ένα πολύ δυνατό πλήγμα. Πέραν λοιπόν των τροπολογιών, πέραν των τροπολογιών ε, όπως η 116 της κυρίας Αγιάλα, η αυτή του κυρίου Γκεμπράντη και άλλων, πρέπει να ενσωματώσουμε τις τροπολογίες αυτές που ουσιαστικά ζητούν νέα διαδικασία υποβολή υποψηφιοτήτων για την θέση του Γενικού Γραμματέα και βέβαια φυσικά την απόσυρση, την παρέτηση του κυρίου Σελμάγερ έτσι ώστε να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία υποβολής προτάσεων και υποψηφιότητων. Μόνο έτσι θα φτάσουμε στον τελικό μας στόχο. Για να μην υπάρχει πλέον από εδώ και πέρα πολιτικοποίηση της θέσης του Γενικού Γραμματέα. Αυτά που έκανε ο πρόεδρος Γιούγκερ από την αρχή της θητείας του και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν πολιτικοποιήσει με έντονο τρόπο αυτήν την θέση. Θα πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουμε με μια νέα διαδικασία έτσι ώστε να σταματήσουμε αυτήν την πάρα πολύ επικίνδυνη διαδικασία ε, πλήγματος αξιοπιστίας που έχει ξεκινήσει. Εγώ πραγματικά, όπως σας είπα, θα υποστηρίξω και τις τροπολογίες του κ. Γκεμπράντη και του κ. Πάστας. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία σας. Μπορώ να πω με πάσα ειλικρίνεια νομίζω ότι, ότι κάποια μέλη του Κοινοβουλίου φοβούνται να έχουν ένα ε, ψήφισμα το οποίο ε, θα ήταν τελώς αποδυναμωμένο, αλλά νομίζω ότι κάνετε εξαιρετική δουλειά, συνεργαστήκατε με το προσωπικό και τη γραμματεία, συντάξατε ένα ψήφισμα το οποίο είναι εύρωστο, αξίζει απόλυτα την ε, υποστήριξή μας και την ευγνωμοσύνη μας. Και νομίζω ότι η θέση σας ε, επεσήμανε περαιτέρω την ακαιρεότητα και την ισχύ αυτής της Επιτροπής και πραγματικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γι' αυτό. Είπατε στη συνεδρίαση ότι τα 4 πέμπτα, το 80% των τροπολογιών που υποβλήθηκαν, θα προτιμούσατε να μην εγκριθούν. Θα βάλετε μείον στον κατάλογο των ψηφοφοριών. Επίσης είπατε ότι θα προτείνετε κάποιες συμβαστικές λύσεις. Ε, περιμένω να τις δω. Αλλά, όσον αφορά τα όσα είπαν όλοι οι προλαλήσαντες, Νομίζω ότι σε αυτό το τμήμα της σημερινής συνεδρίασης θα ήθελα να διευκρινίσω ότι όταν λέμε στην παράγραφο 18 ίσως να αλλάξει και η διατύπωση. Ξέρω ότι έχετε υποβάλει και τροπολογία εσείς η ίδια για τη συγκεκριμένη παράγραφο. Αλλά αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι αυτό που συνέβη θα μπορούσαν αυτοί που βρίσκονται εκτός ευρωπαϊκών οργάνων να θεωρήσουν ότι είναι πραξικόπημα. Κυρία Πρόεδρε, αν όντω αυτή είναι η θέση στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, σίγουρα θα υπάρχουν συνέπειε. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες που λένε ότι το α οδηγεί στο β, που σημαίνει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα. Υπάρχει τροπολογία 116 από τους σοσιαλδημοκράτες, για παράδειγμα, ε, η τροπολογία του κ. Ντεγιούγκ και του υποφαινόμενου και του κ. Γκέρμπραντι και θα ήθελα να πω, κυρία Πρόεδρε, μήπως θα ήταν καλό να κάτσουμε γύρω ένα τραπέζι, οι άνθρωποι που έχουμε υποβάλει τροπολογίε, να βρούμε μια σωστή διατύπωση που θα είναι δίκαιη και θα περιλαμβάνει όλε τι διάφορε εναλλακτικέ λύσει, ενώ ταυτόχρονα θα προτείνει και συγκεκριμένη δράση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και θα επισημαίνει και την πεποίθησή μας ότι αυτό το οποίο συνέβη είναι απαράδεκτο και ότι έχει αμαυρώσει και τη φήμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκκληση λοιπόν που κάνω προς εσάς είναι να μιλήσετε με τα μέλη τα οποία υπέβαλαν τροπολογίες για δράση, έτσι τις αποκαλώ, ε, να τις συζητήσετε για να καταλήξουμε και σε ένα συμβιβασμό που θα αποστέλει ένα σαφές μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ζητά δράση, μεγαλύτερη ε, διαφάνεια και πιο ανοιχτό πνεύμα. Ο κύριος Αλαφράγκα και μετά και πάλι η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι στη συζήτηση που κάνουμε αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι ουσιώδης και πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Η δυνατότητα, τα δικαιώματα και ε, οι δυνατότητες που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον δημοκρατικό έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και νομίζω ότι ως προς αυτό το σημείο δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία. Το θέμα, κυρία Πρόεδρε, είναι πώς ε, ασκούμε αυτό το δικαίωμα δημοκρατικού ελέγχου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά την άποψή μου, αυτό το δικαίωμα το οποίο ε, είναι του Κοινοβουλίου θα πρέπει να ασκείται με υπεύθυνο τρόπο, με αναλογικό τρόπο και με τρόπο ο οποίος θα αρμόζει με την αίσθηση ευθύνης που διαθέτουμε. Εδώ, εσείς κυρία Πρόεδρε, στην εισαγωγή σήμερα και στην αξιολόγηση που κάνετε για τις τροπολογίες, μας είπατε ότι ο στόχος αυτού του ψηφίσματος είναι να ε, είμαστε λίγο διδακτικοί ως προς τη διαδικασία που ακολουθήσαμε και κάποιοι συνάδελφοι, και συμφωνώ με την προσέγγιση αυτή, είπαν ότι θα πρέπει να αντιλήσουμε και κάποια συμπεράσματα από όλη αυτή τη διαδικασία. Η παρουσία εδώ του κυρίου Έτιγκερ διότι εγώ είπα ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη κάποια κριτήρια. Κριτήρια τα οποία δεν αξιολογούνται εδώ, διότι βρισκόμαστε περισσότερο στου τύπου και όχι στην ουσία, είναι η ποιότητα και τα προσόντα του υποψηφίου. Τώρα, ε, το δεύτερο ερώτημα είναι αν η διαδικασία ήταν νόμιμη. Σήμερα η νομική υπηρεσία μας λέει ότι η χρήση του άρθρου 7 μπορεί να οδηγήσει και σε διαφορετικές ερμηνείες. Και σήμερα αυτό το οποίο ήταν απόλυτα σαφές ε, την ημέρα που ήρθε εδώ ο κύριος Έτιγκερ, ε, μετατρέπεται σε διαφορά στην ερμηνεία του άρθρου 7 για να μην χρειαστεί να γίνει διαγωνισμός για την επιλογή προσώπου. Και εδώ, κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Το αν η διαδικασία είναι διαφορετική από αυτή που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο παρελθόν για την επιλογή του Γενικού της Γραμματέα. Και κάτι άλλο το οποίο θεωρώ επίσης ότι είναι σημαντικό είναι τι μπορούμε να κάνουμε συνολικά ως θεσμικά όργανα για το μέλλον, ώστε οι διαδικασίες διορισμών ε, βάσει του κανονισμού να είναι πιο διάφανες διαδικασίες, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις αρχές της αξίας και των ικανοτήτων που εμπνέει ε, το ε, λειτουργήμα του Δημοσίου Υπαλλήλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο ετέθη, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι εμείς δεν θεωρούμε ότι η διατύπωση αυτή, η οποία είναι στεναρή και λέμε ότι πρόκειται περί πραξικοπήματος, είναι αποδεκτή διατύπωση. Για, γιατί κύριε Πρόεδρε, γιατί υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που με ιδιαίτερο στένος υπέβαλαν τροπολογίες με τις οποίες διαφωνώ, λέγοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπεριφέρθηκε με τον ίδιο τρόπο για κάποιους διορισμούς. Και τι σημαίνει αυτό, ότι εμείς ευνοήσαμε ή ανεχτήκαμε πραξικόπημα. Νομίζω, κυρία Πρόεδρε, ότι θα πρέπει να επισημάνουμε εδώ ε, για το μέλλον. Θα μπορούσα να επεκταθώ πολύ περισσότερο, δεν θα το κάνω, για την περιβόητη ιστορία για την ε, νομιμότητα και για τις ε, δυνατότητες να υπάρχουν μεταρρυθμίσεις και τις διαμαρτυρίες, νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στο μέλλον. Θα πρέπει να δεσμευτούμε μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων, ώστε αυτές οι περιπτώσεις να μην επαναληφθούν Κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν κάποιες τροπολογίες οι οποίες υπευλήθησαν που λένε ότι θα πρέπει να σεβόμαστε το γράμμα και το πνεύμα του κανονισμού ε, υπηρεσιακής κατάστασης. Εγώ διαβάζω και στα αγγλικά και στα γαλλικά, αλλά το άρθρο 158 σημείο 1 του κανονισμού μας λέει ότι όλα τα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να διαβιβάζονται και να διανέμονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες. Δεν το λέω ως επίκριση γιατί διαβάζω τέλεια αγγλικά και γαλλικά, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε και λίγο προσεκτικοί για τις ε, συνέπειες που μπορεί να έχουν κάποια πράγματα που λέμε. Παρακολούθησε ιδιαίτερη, με ιδιαίτερη προσοχή την κυρία Γιάλα που μα λέει ότι δεν πρέπει να επιδεινώσουμε την κατάσταση, δεν μπορούμε να οδηγήσουμε σε κρίση. Τι σημαίνει αυτό κυρία Γιάλα, ότι η ε, τροπολογία σας 77 που λέτε ότι αυτό ο διορισμό είναι απαράδεκτο, ε, θα την αποσύρετε, θα μετριάσετε τη θέση σα. Νομίζω ότι ο τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουμε το θέμα αυτό αφορά και την αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια με τη δυνατότητα που έχουμε να ελέγχουμε σε πολιτικό επίπεδο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να το πούμε αυτό, αλλά εγώ δεν θα τολμούσα κυρία Πρόεδρε να πω ότι ήταν παράνομος αυτός ο διορισμός. Γι' αυτά υπάρχουν το δικαστήριο και ε, οτιδήποτε, οποιοςδήποτε θεωρήσει ότι υπήρξε αντικείμενο διάκρισης ή ότι ήταν παράνομη διαδικασία πρέπει να προσφύγει στο δικαστήριο. Εμείς θα πρέπει, και αυτό το είπατε και εσείς κυρία Πρόεδρε και πολύ σωστά, να στραφούμε προς το μέλλον ώστε οι μελλοντικοί διορισμοί να μπορούν να προσαρμοστούν σε κανόνες μεγαλύτερης διαφάνειας και με τρόπο ώστε να λαμβάνουν υπόψη και τις αρχές και τις αξίες και των ικανοτήτων ώστε οι υπάλληλοι να μην νιώθουν ότι ε, τους ε, ε, εμποδίζουν για την επίτευξη των στόχων τους και των προσδικιών τους. Και υπάρχει και κάτι το οποίο πρέπει να ανταποκρίνεται στα γεγονότα. Και εγώ επέβαλα και κάποιες τροπολογίες με τον κύριο Γκονσάλες ε, Πόνς και θεωρούμε ότι είναι πολιτικής φύσεως ε, η διαδικασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή θα σταθούμε σε νομική διαδικασία που επαναλαμβάνω δεν είναι δική μας δουλειά, είναι δουλειά του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ελπίζω, κυρία Πρόεδρε, με την αποδεδειγμένη αντικειμενικότητά σας να υποβάλλετε κάποιες συμβαστικές τροπολογίες και τελικά το κείμενο να αποτελέσει ψήφισμα το οποίο θα υποστηρίξουν οι μεγαλύτερε πολιτικέ ομάδε, χωρί να ξεχνούμε ποιο είναι ο στόχο μα. Που επαναλαμβάνω, δεν είναι να ε, μαλώσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά οι μελλοντικοί διορισμοί να σέβονται τι αρχέ, τι αξίε και τι ικανότητε και να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε ξανά το λόγο. Ήθελα απλώ να σχολιάσω κάτι το οποίο με ανησύχησε και το είπε ο κύριος Ντε τον οποίο σέβομαι απόλυτα για τις θέσεις του και είναι πολύ συνεκτικές και πολύ λογικό, άλλο το αν διαφωνώ ή όχι. Αναφέρεστε σε κάποιους υπαλλήλου που ε, είναι σε διαδικασία να φτάσουν σε βαθμο ld AD15 και τώρα τα της δεν θα το δούμε και θεωρούν ότι διαψεύστηκαν οι προσδοκίε τους. Και αυτό είναι κάτι ακόμα για το οποίο ε, ε, υπέβαλα μια τροπολογία, θεωρείται ότι είναι δευτερεύουσα σημασία, αλλά εγώ θεωρώ ότι έχει μεγάλη σημασία για όλα όσα θέλουμε. Στον κατάλογο που επισυνάπτεται την ημέρα που ελήφθη η απόφαση για τον κύριο Σελμάγερ ε, για γενικό γραμματέα, υπήρχε και ένας ακόμα κατάλογος που είχε μια πολύ σημαντική αλλαγή ε, μεταξύ γενικών διευθυντών. Και αυτό το οποίο με ανησυχεί και χαίρομαι που κάποιοι από αυτούς θα προσφύγουν στο δικαστήριο ε, και χαίρομαι που ελήφθη υπόψη, αλλά θα ήθελα να διευκρινίσουμε και τι δυνατότητα έχουν κάποιοι υψηλά ιστάμενοι αξιωματούχοι για να μην πω πολύ υψηλά ιστάμενοι εξωματούχοι, να ασκούν πιέσει σε κάποια θεσμικά όργανα. Διότι όταν αναφερόμαστε σε άτομα τα οποία τους ε, διακόπηκε η προαγωγή τους σε AD15, εγώ σίγουρα είμαι με τους υπαλλήλου, ε, διότι όταν είναι στη θέση Α14, λογικά μπορούν να πάνε στη θέση AD15 και ξαφνικά βλέπουν κάποια άλλα μέλη ε, του επιτελείου, να μην πηγαίνουν από τον AD14 στο AD15, αλλά ξαφνικά να βρίσκονται εκεί πέρα ε, σε θέση AD15. Και αυτό σίγουρα είναι πρόβλημα και για την απόφαση για τον Γενικό Διευθυντή, αλλά και για την αντίδραση κάποιων ε, υψηλών αξιωματήχων. Εγώ για κάποιους τρία χρόνια ζητούσα αναθεώρηση του κανονισμού, γιατί ήμουνα μέχρι εδώ και δεν ήξερα πώ μπορώ να το αντιμετωπίσω και όχι μόνο εγώ και άλλοι. Εάν λοιπόν φτάσουμε μέχρι εκεί, τότε θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη όλα, γιατί νομίζω ότι και σε αυτή την περίπτωση υπήρχε κάτι περισσότερο και δεν ήταν απλώς ε, τα όσα αφορούν το νέο Γενικό Γραμματέα. Εάν λοιπόν περάσουμε σε αυτό, εγώ συμφωνώ και χαίρομαι που η ε, ομπουτσμαν θα ασχοληθεί με αυτό, αλλά να ασχοληθούμε με όλα, όχι μόνο για το συγκεκριμένο διορισμό, αλλά να τα δούμε όλα από κοινού. Και πώς προχώρησαν αυτές οι δυναμικές. Διότι εδώ αναφερόμαστε στην ανάγκη να υπάρχει ευθύνη για όλους. Και εγώ, και το ξέρω και πολύ καλά, διότι μου ήρθε απευθεία και δεν ε, ε, χρειάστηκε να το ψάξω, γιατί μου φτάνουν εμένα, δεν τα ψάχνω καν, μου έρχονται εμένα. Και ότι αυτό συνέβη. Έλεγα λοιπόν στον κύριο Ντεγιόγκ και στον κύριο Γκερμπράντη και ε, δέχομαι τις προτάσεις ακόμα και αν διαφωνώ εγώ μπορείτε κάλλιστα φυσικά να υποβάλλετε προτάσεις αλλά προσέξτε γιατί σε κάποιες περιπτώσεις νομίζω ότι και εμείς ήμασταν αντικείμενο και στον τύπο σχολιασμών αλλά και γενικότερων σχολιασμών από κάποιους άλλους υψηλά ειστάμενους υπαλλήλους διότι αν κάποιοι φτάνουν ξαφνικά στη θέση 15 θεωρείται ότι έχει την αξία και όταν σου λέει αρμόδια αρχή ότι σε πάβουνε, ε, πας κάπου αλλού, θα διαπραγματευτείς. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διαδικασία για να δούμε και τι γίνεται με αυτούς τους υπαλλήλους, διότι πριν ε, αποσυνδεθούν τα, τα πάντα, θα πρέπει να υπάρχει ένας κατάλληλος διορισμός και μια κατάλληλη διαδικασία για να μην ξαναυπάρξει τέτοια κατάσταση. Και το λέω και με όλη την αγάπη, ε, αλλά εδώ και εβδομάδες ασχολούμαι με αυτό το θέμα ε, ασχολούμαι με το ένα θέμα χωρίς να αγγίζω και το άλλο, το οποίο είναι πολύ μεγάλο τμήμα των επικρίσεων. Θα ήθελα τουλάχιστον να το διευκρινίσω λοιπόν, γιατί εγώ αγαπώ πολύ τους υπαλλήλους, αλλά πιστεύω ότι κάποιοι θα πρέπει να ξαναδούν τον τρόπο με τον οποίο αποδέχονται κάποια πράγματα. Να δέχονται ότι κάποιο όταν φτάσει σε θέση αντί 15, ε, όπου και να πας δεν θα είσαι σε χειρότερη θέση από ό,τι ήσουν και τους γνωρίζω όλους ε, τους υπαλλήλους της Επιτροπής. Ε, σας παρακαλώ λοιπόν λίγο προσοχή. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα θέλει το λόγο. Κύριος Φλάναγκαν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Από αυτά που άκουσα εδώ, ε, βλέπω ότι δεν θα αλλάξουν και πολλά. Ο κύριο Σελμάρη θα παραμείνει στη θέση του, διότι δεν υπάρχει νομική βάση για να τον απομακρύνουμε από αυτή. Θα παραμείνει λοιπόν σε αυτή τη θέση. Δεν θα μπορέσουμε να τον απομακρύνουμε και το σίγουρο είναι ότι αν παραμείνει στη θέση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πληγεί ακόμα περισσότερο. Ναι, αυτό θα γίνει μας έχουν πει πως αυτό ήταν νόμιμο. Όμως ξέρετε κάποια από τα ε, πιο αποτρόπαια εγκλήματα τελέστηκαν ε, υπό το παραπετάσμα της ε, νομιμότητας. Εάν δεν φύγει ο κύριος Σελμάιερ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πληγεί. Αυτό είναι γεγονός και το ξέρουν όλοι, και ο κύριος Γιούνκερ και ο κύριος Σελμάιερ, όλοι. όλα αυτά, επιμένουν και περιμένουν μέχρι να κοπάσει η καταγίδα. Δεν έχει σημασία το τι πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, πώ θα νομίσει το κοινό. Μου φαίνεται πω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ενδιαφέρεται για το τι θα νομίσουν οι πολίτε. Αυτό πλήττει την εικόνα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και επιβεβαιώνει τι υποψίε μου για το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ενδιαφέρεται για το τι σκέφτονται οι πολίτε. Ορισμένοι ε, επίτροποι μάλιστα αποφεύγουν να μας δώσουν τις ε, κατάλληλες απαντήσεις. Η Φεντερίκα Μογκερίνη αποφεύγει επανειλημμένα ε, να απαντήσει για συγκεκριμένα θέματα και ζητάμε απαντήσεις σε ορισμένες ερωτήσεις τις οποίες δεν παίρνουμε ποτέ. Όταν όμως ε, φτάσει ο κόμπος ε, στο χτένι, τότε θα αλλάξουν πολλά. Η ουσία είναι ότι δεν ενδιαφέρεται κανείς για το τι πιστεύουμε και ο κύριος Γιούγκερ θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να επιβεβαιωθεί ο διορισμός του κύριου Σελμάιερ. Και ακούσαμε επίση πως δεν πρέπει να υπερβάλλουμε. Κοιτάξτε, ούτε κι εγώ είμαι ένθερμος υποστηρικτής του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, όμως που είναι υπερβολή εδώ έχει πληγεί η εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το να παραμείνει αυτό το άτομο σε αυτή τη θέση θα επιδεινώσει την κατάσταση. Και αυτό το μπλαζέ ύφο που μας ε, σέρβιρε ο κύριος Σότινγκερ όταν ήρθε εδώ τελευταία φορά ήταν ε, απίστευτο. Σίγουρα, ο διορισμός ήταν πάρα πολύ γρήγορος. Ε, Μα είπε ο κύριο Σέτινγκερ ότι η διαδικασία διορισμού ε, κράτησε έξι εβδομάδες, αλλά δεν υπήρξε καμία υποστήριξη με επιχειρήματα. Τι θα γίνει όμως στην περίπτωση που ας πούμε ο κύριος Σέτινγκερ αρρωστήσει για ένα διάστημα τεσσάρων ή έξι εβδομάδων, αν πιστέψουμε τα λόγια του, καταστροφή. Θα διαλυθούν τα, τα πάντα. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, είπε ο κύριο Σότινγκερ. Όχι, ο κύριο Σελμαΐρ. Άλλο ο κύριο Σελμαΐρ, αρρωστήσει και λείψει για 6 εβδομάδε, τι θα γίνει, θα διαλυθεί η Κομισιόν. Αυτό που ακούσαμε στην ουσία ήταν ότι ένα από του λόγου που πήρε ο κύριο Σελμάρη αυτή τη θέση ήταν ότι δεν μπορούσαμε να περιμένουμε όλον αυτό τον καιρό που χρειαζόταν μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ναι, και θα το ξαναπώ, το θα το ξαναπώ. Πώς, γίνεται να υπερβάλλουμε σε αυτή την περίπτωση. Αυτό που συνέβη ήταν ε, καταστροφή. Και πιστεύω ότι ο κύριος Κερμπράντι είπε ε, το σημαντικότερο που ακούσαμε σήμερα. Ούτε καν παραδέχτηκε κανένας από την Κομισιόν ότι η διαδικασία ήταν προβληματική. Εμείς λοιπόν μπορούμε να ψηφίσουμε αυτό το κείμενο εδώ, αλλά εάν έστω και ένας ευρωβουλευτής υπερψηφίσει, παραμένει σε αυτή τη θέση που μας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, εκούσια πλήττει την εικόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τι μας λέει αυτό? Σίγουρα τίποτα καλό. Δεν μπορούμε να υπερβάλλουμε. Δεν υπάρχει δυνατότητα να υπερβάλλουμε για κάτι τέτοιο. Αυτό είναι απίστευτο. Also... Μάλιστα. Θα Ήθελα και εγώ να κάνω κάποια σχόλια, κάποιες παρατηρήσεις πάνω στην όλη συζήτηση. Να πω, τι ήθελα να πω πριν πάλι στα πάρει το λόγο ο κύριος Φλάνναγκαν, ότι ε, με ικανοποίησε πάρα πολύ η αντικειμενικότητα και ουδετερότητα αυτή τη συζήτηση, όμως μετά πήρε το λόγο ο κύριος Φλάνναγκαν. Ε, συνάδελφε, κύριε Κλίντς, ζητήστε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για μένα η κατάσταση έχει ως εξής. Υπάρχουν τρεις πτυχές σε αυτό το θέμα. Υπάρχει η νομική πτυχή, υπάρχει η διαδικαστική ε, πτυχή για τις ε, αρμοδιότητες και για και οι αρμοδιότητες μάλλον. Τώρα, πώς μου φαίνονται μένα τα πράγματα. Νομίζω πως όλα είναι θέμα οπτικής γωνίας. Ε, σίγουρα υπάρχουν θέματα διαφάνειας, αλλά κάποιος άλλος μπορεί να ισχυριστεί ότι όλα έγιναν σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Οι συνάδελφοι πριν από μένα μίλησαν για ένα άνευ προηγουμένου σκάνδαλο, το οποίο θα ε, κατακριμνήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια βαθύτατη κρίση, αν παραμείνει στη θέση αυτή ο κύριος Ελμάιερ. Τώρα, το ότι το θέμα αυτό είναι αμφιλεγόμενο δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά οποιοδήποτε ανώτερος υπάλληλο, αν είχε την ευκαιρία να ανελιχθεί τόσο γρήγορα, θα θα έλεγε όχι. Αυτό είναι σίγουρο. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο κύριος Γιούγκερ, ήταν υπέρ ενός τέτοιου διορισμού και σίγουρα δεν ήταν ο μόνος, δεν ενήργησε αυθαίρετα. Τώρα, αν θέλουμε να κάνουμε τον κύριο Σελμάιερ μαύρο πρόβατο ή αποδιοποπέο τράγο, εντάξει, μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά αυτό δεν ε, δείχνει ότι φταίει ο κύριος Σελμαίερ. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα ίσως ε, στον ε, κανονισμό. Επίσης, θεωρώ πως το θέμα των αρμοδιοτήτων δεν έχει αμφιλεγόμενα σημεία, δεν έγινε κάτι παράτυπο. Ο κύριος Σελμάιερ σίγουρα δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν είναι κατάλληλος για το πόστο αυτό. Το αντίθετο μάλιστα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ε, είναι πάρα πολύ ικανός, το έχει αποδείξει αυτό και μπορεί να αναλάβει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το να ζητήσουμε την ανάκληση του διορισμού του κυρίου ε, όπως είπε και Ισπανός συνάδελφος, ε, διότι πρόκειται περί εγκληματικού διορισμού κτλ. Αυτά για μένα είναι πολύ βαριά λόγια. Δεν έχουν θέση σε ένα ψήφισμα. Το αντίθετο, αυτό που θα έπρεπε να, να ε, κάνουμε είναι να είμαστε πιο ήπιοι στις εκφράσεις μας και να φροντίσουμε να μην πληγεί ακόμα περισσότερο η ε, φήμη και εικόνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε να ανακληθεί ο διορισμός ενός ατόμου το οποίο πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και έχει όλα τα προσώτα να αναλάβει αυτά τα καθήκοντα. Και επίσης, ο αναμάρτητος πρώτο στο λιθοφαλέτο, Ξέρετε τι λένε. Και εδώ αν ψάξουν μπορούν να βρουν διάφορες ε, περιπτώσεις όπου δεν ε, υπήρχε απόλυτη διαφάνεια. Όχι μόνο εδώ αλλά και ε, στα κρατημέλη και σε διάφορους εθνικούς διορισμούς. Θέλετε να αρχίσουμε λοιπόν αυτές τις διαδικασίες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τώρα όλους που λάβατε το λόγο. Θα προσπαθήσω να συνοψίσω και να πω ότι ότι ακούσαμε Ακούσαμε τις απόψεις και πάνω κάτω υπάρχουν 40 ψήφοι υπέρ και 19 ψήφοι κατά του ψηφίσματος. Εδώ αυτό δείχνει για μένα ότι έγινε μια βαθύτατη ανταλλαγή απόψεων και γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους, διότι ακούσαμε όλες τις απόψεις τοποθετηθήκατε όλοι πάνω στις ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σίγουρα δεν ε, μπορεί να συμφωνούμε όλοι με αυτά που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ακριβώς αυτή η πληθώρα απόψεων μας δείχνει τη δημοκρατικότητα της ε, διαδικασίας. Σίγουρα δεν μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε και πρέπει να βρεθεί μια μέση λύση η οποία θα συμπεριλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία από τις απόψεις των ε, περισσότερων. Αυτό που με λυπεί περισσότερο είναι η πίεση χρόνου που έχουμε υπόστη για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Δεν είχαμε καθόλου ε, πολύ χρόνο στη διάθεσή μας για να εντοπίσουμε ε, τα προβληματικά θέματα, για να καταρτήσουμε έναν κατάλογο με ερωτήσεις ε, με επίμαχα σημεία. Μετά έπρεπε πολύ γρήγορα να περάσει όλο το κείμενο στη σειρά των ε, νομικών υπηρεσιών για να το ελέγξουν. Λυπάμαι λοιπόν πάρα πολύ για την έλλειψη χρόνου που είχαμε και το είπε και ο κύριος Αλαφράγκα ε, για την παράγραφο 18 ότι για αυτούς τους λόγους είναι προβληματική. Και αυτή η έκφραση το could be seen as δικαιολογείται στο ψήφισμα αυτό ακριβώς για να αντικατοπτρίζεται όλο το εύρος των απόψεων. Βέβαια το considered είναι και αυτό μια καλή πρόταση που είπε ο συνάδελφος. Ε, πιστεύω πως πρέπει ε, πάση θυσία να αντικατοπτρίζεται αυτό το εύρος των απόψεων στο ψήφισμα. Μετά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι λοιπές το ψήφισμα, ότι πρέπει να πούμε και άλλα, να γίνουν και άλλα να πω εδώ στον ε, κύριο Ντεγιόν ότι δεν ε, διεκπεραιώνουμε το θέμα και περνάμε παραπέρα. Οι σοσιαλδημοκράτες ε, μπορούν να συνεχίσουν να υποβάλουν προτάσεις. Το θέμα είναι τι κάνουμε στο μέλλον. Και εδώ δίνω τη σκητάλη σε εσά και να πω ξανά ότι σα ευχαριστώ για αυτήν την συμμετοχή στην ανταλλαγή απόψεων. Έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα και πρέπει να ε, δουλέψουμε έτσι ώστε να μην χρειαστεί και του χρόνου να ξαναπιάσουμε το θέμα αυτό από την αρχή. Και είναι ένα θέμα το οποίο εντοπίσαμε, είναι ένα θέμα το για το οποίο συμφωνήσαμε πώς δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να περάσει ε, έτσι, χωρίς αντίδραση. Πρέπει επίσης να απαντήσουμε στο ερώτημα ε, ποιον ακριβώς θέλουμε σε τέτοια υψηλά πόστα. Θέλουμε υπαλλήλου ε, καριέρας, θέλουμε πολιτικούς διορτισμούς, τι δεν θέλουμε. Αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να συζητηθούν σύντομα και ο εσωτερικός κανονισμός κάθε φορά που τίθεται επί διάταξη διάταξης αυτήν εδώ την Επιτροπή μας οδηγεί σε μεγάλες συζητήσεις, διαφωνίες, τσακωμού. Το έχετε δει πάρα πολλές φορές. Κάθε φορά που ασχολούμαστε με τον εσωτερικό κανονισμό. Φτάνει πια. Δεν πρέπει να επαναλαμβάνονται αυτές οι συζητήσεις. Δεν βοηθά κανέναν. Νομίζω πως η πρόταση του κυρίου Ότινιερ δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητη. Πρέπει να την εξετάσουμε και πρέπει να την πάρουμε στα σοβαρά. Μέχρι τώρα έχουμε δει ότι κάθε προσπάθεια ε, που κατέβαλε η Επιτροπή για την ε, αλλαγή του κανονισμού δεν οδήγησε πουθενά. Αυτός ο κανονισμός ε, της Κομισιόν για το προσωπικό έχει έχει λήξει μέχρι το 2020, το αργότερο μέχρι το 2023. Πρέπει λοιπόν να το πάρουμε στα σοβαρά το θέμα αυτό. Τώρα, αυτό σας το υπόσχομαι, ότι δεν θα παραπέσει. Και να είστε σίγουροι πόσο πολλοί έχουν τα βλέμματα στραμμένα στις Βρυξέλλες και παρακολουθούν τις εξελίξεις και πρέπει τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να διαλευκάνουμε ορισμένα σκοτεινά σημεία. Σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Υπάρχουν προβλήματα και τα προβλήματα που υπάρχουν όμως δεν πρέπει να αποσιωπούνται, πρέπει να συζητηθούν. Και να πω τώρα κάτι προσωπικά στον κύριο Γκεμπράντη. Οι δικές σας τροπολογίες που αναφέρονται στην διαμεσολαβήτρια ε, να σας πω πως δεν είμαι σίγουρη για το αν πρέπει να χρησιμοποιούμε τόσο έντονα λόγια, να μην είμαστε τόσο απόλυτοι, άσχετα από το τι θα συμβεί. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να είστε πιο προσεκτικοί στην ε, διατύπωση ε, των τροπολογιών σας σχετικά με την ε, ανάκληση του διορισμού του Γενικού Γραμματέα. Δεν μπορούμε να πετήσουμε από το Σώμα των Επιτρόπων τρεις εβδομάδες αργότερα να αλλάξει γνώμη και να πάρει πίσω μια απόφαση. Εάν γίνει επίκληση στο άρθρο 15 και στη χρυσή χειραψία, όπως λέγεται, τότε θα υπάρξουν προβλήματα. Και εγώ διαφωνώ γι' αυτό. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνω ότι πρέπει να αποφύγουμε τις αναφορές σε ανάκληση του διορισμού. Πρέπει να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο αντικειμενικοί. Και σίγουρα δεν είναι κάτι το οποίο είναι ευχάριστο για κανέναν από εμά, όμως χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Όλες λοιπόν αυτές οι τροπολογίες θα εξεταστούν, θα ξαναμιλήσουμε και με τον ε, συνάδελφο Στάς. Την Τετάρτη βέβαια, γιατί δυστυχώς ε, αύριο πρέπει να πάω στη Στουγκάρτη, γιατί έχουμε διάφορα θέματα εκεί διοικητικά. Την Τετάρτη λοιπόν θα επιστρέψω και θέλω να συζητήσω με τον κύριο Στάση, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αν θα καταφέρουμε να έχουμε μια πλειοψηφία για ε, το, για την ψηφοφορία της ερχόμενης εβδομάδας. Δεν πιστεύω πως χρειάζεται να επιδεινώσουμε και να, τα πράγματα, να οξύνουμε την κατάσταση. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσεκτικός λόγος στο ψήφισμα. Όμως, επαναλαμβάνω, θα συζητήσουμε και με την γραμματεία, θα τα δούμε όλα πάρα πολύ προσεκτικά στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Νομίζω πως ε, όλο αυτό το θέμα έχει πολλές πτυχές και πολλαπλές επιπτώσεις. Σίγουρα τα κράτη-μέλη δεν θέλουν συγκέντρωση εξουσίας, δεν θέλουν να αποδυναμωθεί ο δικός τους ρόλος. Και δεδομένων όλων αυτών πρέπει και εμείς να αναλογιστούμε τι θέλουμε να καταφέρουμε. Θέλουμε να είμαστε ένας πραγματικός σημαντικός εταίρος της Κομισιόν έτσι ώστε να πάμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα πιο μπροστά. Δεν προσπαθώ να σας πείσω για κάτι. Αναφέρομαι στην ενότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρομαι και στην ενότητα εντός του, της δικής μου πολιτικής ομάδας. Πρέπει να πασχίζουμε για τη βελτίωση, τη βελτίωση σε όλους τους τομείς της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο δημοσιονομικό και ε, στον εσωτερικό διότι αν δεν ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο θα σκοντάψουμε στον επόμενο. Και χρειάζεται επιτέλους πυγμή έτσι ώστε να ληφθούν αποφάσεις οι οποίες θα εφαρμοστούν. Δεν ωφελεί κανένα να σκοντάφτουμε κάθε λίγο σε νέα προβλήματα. Αυτό ας μην το ξεχάσουμε. Αυτά όσον αφορά τις παρατηρήσεις από μένα. Αν έχει κάποιος ένα τελευταίο σχόλιο, παρακαλώ να το κάνει τώρα. Ναι, να πω απλώς ότι καταλαβαίνω ότι το να ανοίξουμε τους κανόνες του προσωπικού, του κανονισμού υπηρεσιακή κατάστασης είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Αλλά υπάρχει κάτι το οποίο έχει σχέση με τον εσωτερικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι και η ανακοίνωση του ε, Πρόεδρου Γιουνκέρ για τα επιτελεία τους ε, ε, να ξέρουν δηλαδή καλύτερα και το προσωπικό ότι υπάρχουν τρόποι να γίνουν κάποια πράγματα ότι αυτά δεν μπορεί να γενικευθούν και κάθε πέντε χρόνια ξέρουμε πώς αλλάζει τα πράγματα και περισσότεροι ασχολούνται με αυτό και όχι με αυτό που θα έπρεπε να τους απασχολεί. Αυτό λοιπόν θα πρέπει ε, κάπως να αλλάξει. Υπάρχουν πιο ήπιοι κανόνες που είναι ο εσωτερικός τρόπος να αλλάζουν τα χαρτιά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ αναγνωρίζω και την αξία των ανθρώπων που εργάζονται στα επιτελεία των Επιτρόπων. Δεν θέλω ούτε να τους στήξω, ούτε να τους μεώσω τα κίνητρα, αλλά έχουμε όλοι προσωπικό παντού για να μπορέσουμε να βρούμε αρκετά άτομα ε, με ε, προσόντα και να τους δώσουμε και κίνητρα να εργαστούν στο επιταλείο των επιτρόπων, αλλά όχι εις βάρος του υπολείπου προσωπικού, διότι έτσι χάνεται όλη η αξιοπιστία και πιστεύω και ο Γενικό Διευθυντή είπε και εσύ ότι πρέπει να είναι κάποιο ο οποίο τα χέρια τη εμπιστοσύνη του Προέδρου για να είναι ισχυρό. Ναι, μεν, αλλά με τον τρόπο αυτό που βρήκαν ε, τελικά ε, δεν θα λειτουργήσει το σύστημα. Εγώ Απλώ πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει με άλλο τρόπο και σε διαβεβαιώνω ότι δεν θα γίνει αυτό, γιατί αυτό το οποίο δημιουργήθηκε δεν το δημιουργήσαμε εμεί και πρέπει και εμεί να συνειδητοποιήσουμε ότι αν στείλει ένα ισχυρό μήνυμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι απαραίτητο διότι το χρειαζόμαστε όλοι για να μπορέσουμε να εμπιστευτούμε και την Επιτροπή και το Γενικό της Γραμματέα. Εννοείται ότι από την τελευταία φορά που υπήρξε το 2014 αναθεώρηση του κανονισμού έχουν ε, έτσι και αλλιώ και εδώ αναφέρομαι στο άρθρο 12, αλλάξει οι κανόνες ε, για όλες τις θέσεις, κυρίως τις ε, διευθυντικέ θέσεις. Υπάρχουν νέοι κανόνες, νέε απαιτήσει. Είναι σαφές ότι αν πάμε στις πιο πάνω θέσεις και αν θες λύσουμε πραγματικά να υπάρξει η δυνατότητα κάποιος εξωτερικός να αναλάβει μια τέτοια θέση θα πρέπει να ξαναδούμε πολύ προσεκτικά ε, αυτό που εσείς ονομάζετε επιβολή ή ε, αλεξιπτοτιστής ο οποίος επιβάλλεται εκ των άλλων θα πρέπει να δούμε πώς θα διευθετηθεί γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχει δυνατότητα και μιας ε, εξωτερικής αν θέλετε στελέχωσης είναι ένα θέμα που σίγουρα θα πρέπει να το επεξεργαστούμε και βέβαια κανείς από μας δεν ε, ασχολείται ευχάριστα με το θέμα αυτό, ιδιαίτερα όταν αφορά το δικό μας θεσμικό όργανο. Ναι, ο κύριος Αλαφράγκα. Κυρία Πρόεδρε, δεν θέλω τώρα να περιπλέξω περισσότερα τα πράγματα, ούτε τα παρατείνω τη συζήτηση. Συμφωνώ με αυτό που λέτε και ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε και μια συνένεση που θα λάβει υπόψη όλες τις ευαισθησίες και κυρίως ε, τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως ε, όργανο το οποίο ελέγχει πολιτικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μία παρατήρηση που έκανε και η κυρία Γιάλα και με την οποία συμφωνώ, διότι πολλές φορές οι υπάλληλοι θεωρούν ότι ε, δεν έχουν δυνατότητες προαγωγής, αλλά αυτά τα οποία λέμε για τα επιτελεία των επιτρόπων και είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη για τα επιτελεία όλων των θεσμικών οργάνων. Και γνωρίζουμε όλοι ε, ποιες είναι οι προνομιακέ θέσει, επί τη βάση βέβαια τη αξία, γιατί αναλαμβάνουν πάρα πολύ καθήκοντα τα άτομα τα οποία εργάζονται στα επιτελεία, αλλά είναι ε, μια γενικότερη παρατήρηση που αφορά το Γενικό Γραμματέα σε αυτή την περίπτωση, αλλά σε άλλε περιπτώσει αφορούσε και γενικού διευθυντέ, ε, ε, υψηλά ειστάμενου αξιωματούχου των θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ολοκληρώσαμε το σημείο αυτό στην ημερήσια διάθεση για τα διάφορα. Δεν υπάρχει κανεί στον υποβολή Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη δημόσια συζήτηση και θα ακολουθήσει μια πολύ σύντομη συνάντηση των συντονιστών. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ για την παρουσία όλων.